Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Ε. ε. είναι διαδικαστικό το θέμα που θέλετε να θέσετε. Mr. President. Πρόεδρε. Και πάλι θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για, το για τη διαχείριση του χρόνου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χτες και σήμερα ε, καταπατήσαμε το χρόνο ε, που προβλεπόταν για την ε, ψηφοφορία. Μα πρέπει να δίνουμε την εικόνα ενό κοινοβουλίου που λειτουργεί εύρυθμα, που διαχειρίζεται σωστά το χρόνο. Μπορείτε σας παρακαλώ να αποταθείτε στις αρμόδιες αρχές γιατί αλλιώς θα μας περιφρονούν και θα το αξίζουμε αν συνεχίσουμε έτσι. Go ahead. Go ahead. Παρακαλώ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, το δικό μου το διαδικαστικό αφορά τις ε, δύο πρώτες ε, ψηφορίε που έχουμε για το χονδιάγραμμα το περίοδο συνόδου του 12 και του 13 και έχω εδώ να θίξω δύο θέματα. Πρώτον, αυτέ οι δύο ψηφορίε απλά καταδεικνύουν πόσο αδύναμο είναι στην ουσία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι μιλάνε για μεγαλύτερη δύναμη και εξουσία, αλλά επί τη ουσία, σας παρακαλώ λέει ο πρόεδρο. κύριε Κλάρκ, ε, διαδικαστικό, όχι ομιλία. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι είμαστε δεσμευμένοι. Κλείνει το μικρόφωνο ο λοιπόν πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην ψηφορία και αφαιρεί το λόγο από τον ομιλητή. As Όπως ξέρετε συνάδελφοι, ε, θα, μετά την ε, ομιλία του Πρόεδρου της Ουγγαρίας, του κυρίου Σμίτ, θα ψηφίσουμε για το χρονοδιάγραμμα των περίοδων συνόδου του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ. Πρόεδρε, Υπό ε, συνθήκες ε, δεν θα ζητούσα το λόγο για να ε, παρέμβω, διότι σέβομαι τον Πρόεδρο, γιατί και εγώ Πρόεδρος είμαι. Ε, όμως, όμως έμαθαν τα πολιτικά κόμματα ότι υπάρχουν τροπολογίες που θα συζητηθούν πριν την ψηφοφορία και όχι μετά την ομιλία του Πρόεδρου της Ουγγαρίας. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό στον κύριο Σμιτ. Δηλαδή θα πρέπει να αποχωρήσουν όλοι και να επανέλθουν για τη δεύτερη ψηφοφορία. Σα προτείνω λοιπόν να τροποποιήσουμε την ημερήσια διάταξη, ούτω ώστε όλε οι ψηφοφορίε να έχουν ολοκληρωθεί πριν την ομιλία και να ξεκινήσουμε μάλιστα με την ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα. Uh, Mr. Mr. Κύριε Μακμίλαν Σκότ, ε, μπορώ να σας απαντήσω σε αυτά που είπατε με την εξή έννοια ότι τη Δευτέρα το Κοινοβούλιο ψήφισε για την ημερήσια διάταξη της Συνόδου αυτής και εκεί βλέπετε το Κοινοβούλιο ενέκρινε η ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα να γίνει ε, την ώρα που αναφέρεται εδώ στην ημερήσια διάταξη. Άρα δηλαδή είναι ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή που αναφέρεται. Ε, κύριος Μακμίλεν Σκοτ. Ε, ζητώ συγγνώμη που καθυστερώ, αλλά οι ε, κατάλογοι ψηφοφοριών μοιράστηκαν σε όλες τις πολιτικές ομάδες και αν αυτό είναι λάθος πρέπει να διορθωθεί. Είναι γελίο και είναι και έλλειψη σεβασμού προς ένα πρωθυπουργό να μας καλέσετε εδώ και πάλι μετά την ομιλία του. Ας το κάνουμε λοιπόν όπως προβλέπετε στον κατάλογο των ψηφοριών και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αλλαγή που έγινε.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 Λοιπόν, ακούστε πώς ε, θα ε, εξελιχθούν, ε, θα διεξαχθούν οι ψηφοφορίες. Μάλλον, ακούστε τι προβλέπετε από τον κανονισμό. Συγγνώμη, μην με αποδοκιμάζετε έτσι. Αν θέλετε να τροποποιήσουμε το καταστατικό. Τι Δευτέρε αποφασίζουμε το χρονοδιάγραμμα για τις ψηφοφορίες. Οι βουλευτέ το αποφάσισαν. Παρ' όλα αυτά, έχει το δικαίωμα ο πρόεδρο να θέσει και πάλι το πρόγραμμα της Ολομέλειας σε ψηφοφορία επιθυμείτε. Χρησιμοποιώ αυτή τη διακριτική ευχαίρεια που έχω και σα ρωτώ, θέλετε να τροποποιήσετε την σειρά των ε, ψηφοφορίων. Ποιο είναι υπέρ του να τροποποιήσουμε ε, το πρόγραμμα. Κατά ε, αποχέ, πάρα πολύ ωραία. Having said this, dear colleagues... Τούτου λεχθέντος σας ε, ε, υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να είστε εδώ τη Δευτέρα αν θέλετε να ακούγεται η άποψή σας και να λαμβάνετε υπόψη σχετικά με τον προγραμματισμό των εργασιών της Ολομέλειας. Ποια ήταν η πρόταση του κυρίου Μακμίλαν Σκοτ. Να ε, προβούμε στην ψηφοφορία για το χρονοδιάγραμμα πριν από την ομιλία του Προέδρου της Ουγγαρίας εάν έχουμε χρόνο. Βλέπετε ότι με όλα αυτά χάνουμε και χρόνο. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει ούτω ή άλλω να συνεχίσουμε μετά την ομιλία, γιατί έχουμε πάρα πολλέ ψηφοφορίε. Ποιο είναι υπέρ του να ψηφίσουμε για το χρονοδιάγραμμα πριν την ομιλία του Προέδρου τη Ουγγαρία, αν μα το επιτρέψει και ο χρόνο. Κατά παρακαλώ. Αποχέ. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Θα ψηφίσουμε για το χρονοδιάγραμμα εάν έχουμε χρόνο πριν την ομιλία ε, του Προέδρου της Ουγγαρίας. Makes no difference. We will anyway vote after. Συνάδελφοι, ούτως ή άλλως θα συνεχίσουν οι ψηφοφορίες μετά την ομιλία του κυρίου Σμιτ. Okay. Πρόεδρος, να σας πω λοιπόν τι θα κάνω. Θα καταφύγω στην προνομία που έχω και για να σταματήσει αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα, ψηφίζουμε τώρα. Πρώτη ψηφορία για το χρονοδιάγραμμα. Συμφωνείτε όλοι, θαυμάσια. Ξεχνάτε ότι είστε και μετά την ομιλία του Πρόεδρου εδώ για να ψηφίσετε, αλλά ας ξεκινήσουμε. Χρονοδιάγραμμα λοιπόν του 2012, ε, τροπολογία 2. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 θα τεθεί σε ψηφοφορία με μυστική ψηφοφορία. Που θα πει θα δείτε το μπλε φωτάκι μπροστά σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία επί του των περιόδων για το 2013. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 με μυστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Έκθεση Φερνάντες, κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προπολογισμού 2012. Τροπολογία Uh, Φοβάμαι, λέει ο Πρόεδρος, ότι σας έδωσα την εντύπωση ότι τελικά η ψηφορία ε, θα μετατραπεί σε καρναβάλι, σε τσίρκο. Η τροπολογία διαπορρίπτεται, η απόφασή μου παραμένει. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 13 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Check. Amendment 2. Check. Τροπολογία 2 ελέγχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, η παράγραφος 31 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας οφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Με συγχωρείτε. Uh, Α, η τροπολογία 7 απεσύρθη. Επομένω, τροπολογία... I'm sorry. Okay. Τροπολογία 7 δεν υπάρχει πλέον ε, δεν υπάρχουν δύο μέρη. Όλοι οι επτά. Ποιοι είναι υπέρ της επτά. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. Check 7. Έλεγχος για την επτά. Πέρα οφορίας. Εγκρίν. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Τσεκ. Τσεκ τροπολογία 1. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η τελική ψήφος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Φερνάντες. Η μερίσια διάσταση προβλέπει ψηφοφορία στην πρόταση ψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Check. Amendment 1. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψήφος με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα της Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Αγαπητοί συνάδελφοι, διακόπτουμε για την ομιλία του Πρόεδρου της Ουγγαρίας και επιστρέφουμε μετά.